Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω τη συνεδρίαση γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε και όταν φτάσουμε στην έκθεση του κυρίου Μπόνη και στην ψηφοφορία θα έχουν έρθει όλοι. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσουμε γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει κατά 6 λεπτά. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ερχόμαστε τώρα στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Το γλωσσικό καθεστώς το γνωρίζετε. Έχουμε τερμηνία στα δανέζικα, θα έχουμε τερμηνία στα δανέζικα, μαλτέζικα, γαελική και ουγγρικά. Και έχουμε τώρα τον, τον ορισμό των εισηγητών. Ο πρόεδρος, κ. Μωράης, έχει οριστεί εισηγητής στο, ε, για, το, για το σχέδιο εφαρμοστικής απόφασης του Συμβουλίου που θα εγκρίνει τα συμπεράσματα της Ευρωπόλ για τη συμφωνία ε, για την συνεργασία μεταξύ Γεωργίας και Ευρωπόλ. Ο κύριος Μπόνι έχει οριστεί εισηγητής για την ανταλλαγή πληροφοριών για τα συστήματα εγκαίρης προειδοποίησης και για την διαδικασία ανάλυσης κινδύνου για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες. η κυρία Μακόβεϊ θα αναλάβει την έκθεση ε, για την Eurodac και τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων και την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού 604. Να σας πω ότι ο προηγούμενος εισηγητής έχει αποσυρθεί, ο κύριος Χοπ και ο κύριος Ντάλτον θα αναλάβει την έκθεση ανταλλαγή πληροφοριών με υπηκόους τρίτων χωρών στο έκρηση. Είναι η έκθεση έκρηση για το, σύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τα αρχεία ποινικών δεδομένων. Η κυρία Βερσιά είναι η για ε, τις κινήσεις προσφύγονται και μεταναστών, το ρόλο του, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή στηρίζει αυτές ε, τις συστάσεις, αυτές τις προτάσεις. Εάν ναι, έχω άλλες δύο ανακοινώσεις να κάνω, να έχετε τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να τις έχετε έτοιμες και από ό,τι κατάλαβα έχουμε και γερμανικό τηλεοπτικό συνεργείο το οποίο είναι παρόν. Προσύμπεν, νομίζω ε, λέγεται ο σταθμός, εκτός και αν το προφέρω λάθος, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά εάν συμφωνείτε όλοι θα παρίσταται το γερμανικό τηλεοπτικό συνεργείο. Πάμε λοιπόν ε, στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης τους κανόνες αστικού, ε, αστικού δικαίου για τη ρομποτική. Η είναι ο κύριος Μπόνι. Κύριε Μπόνη, θα μας, θα μας παρουσιάσει ο κύριος Μπόνη σήμερα ε, το σχέδιο γνωμοδότησης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ασχολείται με την έκθεση για τους κανόνες αστικού δικαίου για τη ρομποτική και η δική μας Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών συντάσσει γνωμοδότηση βάση, βάση του 54. Η ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνικής, τεχνητής νοημοσύνης θα φέρει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία μας, παρόλο που υπάρχουν ανησυχίες και απειλές. Από πλευράς Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών έχω προετοιμάσει ένα σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο εστιάζει την προσοχή του στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την ανάπτυξη των ρομπότ και των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Μέρος της νομοδότησης το έχω αφιερώσει στις δεοντολογικές πτυχές ε, του θέματος, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι αρχές του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να ε, ισχύσουν από την έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού αυτής της τεχνολογίας. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερως η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Ζητούμε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον να περιλάβει διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και αρχές που θα γίνουν γίνονται σεβαστές και που θα τηρούν την ιδιωτικότητα και ότι αυτό θα είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση ήδη από τον σχεδιασμό των ρομπότ. Και σε κάθε περίπτωση η τεχνολογία ε, τεχνητής νοημοσύνης και ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιείται με πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Μας ενδιαφέρει το θέμα της ασφάλειας των συστημάτων και της ροής των δεδομένων. Είναι σημαντικό ε, διότι τα ρομπότ θα αλληλεπιδρούν και θα συνδέονται με διάφορες άλλες συσκευέ. και θα πρέπει τα, προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτικότητα να προστατεύονται. Το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα φωνητικής αναγνώρισης που θα είναι καθοριστικά για την επικοινωνία ανθρώπων και ε, ρομπότ. Και έχω και μία αναφορά στα μη επανδρομένα αεροσκάφη που αντικατοπτρίζει την άποψη της ε, Επιτροπής μας έτσι όπως την εγκρίναμε στην περσινή γνωμοδότηση. Και έχω περιλάβει και ε, την κατάρτιση δεντολογικών κατευθυντηρίων γραμμών για το θέμα της ε, ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό στη γνωμοδότηση γιατί αναφέρεται στα προβλήματα που οι σχεδιαστές και οι χειριστές των ρομπότ θα αντιμετωπίσουν, θα αντιμετωπίζουν μάλλον καθημερινά. Επομένως είναι καλύτερο να υπάρχει ε, δεντολογικός κώδικας το συντομότερο δυνατόν για να μην υπάρξουν παρανοήσεις και για να μην υφίστανται οι σχεδιαστές και οι όλη αυτή την επίεση ε, ξαφνικής υπερβολικής νομοθέτησης. Χρειαζόμαστε κανόνες εξ αρχής και μάλιστα ισχυρούς. Καταληκτική προθεσμία τροπολογιών 11 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνιακή ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Θα λάβει χώρα το αργότερο στις 17 Νοεμβρίου. Ζητώ από τον Πρόεδρο να κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε την ψηφοφορία νωρίτερα γιατί η Επιτροπή Γιούρι ψηφίζει ε, την έκθεση ε, στα τέλη Νοεμβρίου και θα ήταν καλό οι νομοδοτήσεις των λοιπόν κοινοβουλευτικών επιτροπών να είναι έτοιμες. Έπρεπε να είχα πει ότι η Γιούρι είναι καθήλυν αρμόδια, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές στους ε, συντονιστές. Έχουμε και άλλα θέματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων ε, τα συζητήσαμε και θα τα ξανασυζητήσουμε. Και σημειώνω επίση ότι η ημερομηνία προθεσμία υποβολής υποβολή τροπολογιών δεκάτη του μηνό. Ε, θέλει κανείς το λόγο, κύριε έτσι Δράτω με τι ευκαιρίες για να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για το έργο του το σχέδιο είναι ισορροπημένο, σύμφωνα με τις περισσότερες πτυχές του. Αναγνωρίζουμε τις τελευταίες εξελίξεις τη ρομποτική και την τεχνική νοημοσύνη. Τα σχόλια αφορούν ακριβώς τις ε, επικοδομητικές χρήσεις αυτών των τεχνολογιών. Η ρομποτική σε ορισμένε περιπτώσει αξιοποιείται στον τομέα τη υγεία. Επισκέφθηκε ένα τέτοιο σχετικό κέντρο όπου συνεχάριν του προτεργάτε. Πρέπει όμω η χρήση να υπόκειται σε κανόνε ηθική, δεοντολογία και προστασία των ανθρώπων, προστασία επίση των προσωπικών δεδομένων. Η τεχνολογία λοιπόν πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο επικοδομητικό στην υπηρεσία τη κοινωνία, Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία προείπε ο εισηγητής. Η πρόταση στην τεχνολογία, στην ιατρική, στις μεθόδους διάσωση, πρέπει να αποτελούν δρόμους στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μπροστά. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν στην έρευνα, στην καινοτομία, όμω όλα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να αξιοποιούνται για πολεμικές εφαρμογές. Επίσης, δεν πρέπει ο... η χρηματοδότηση να δείτε σε συστήματα διτής χρήσης. Έχουμε και τροπολογίες. Θα τις υποβάλλουμε και για μια φορά συγχαρητήρια θα έχετε κύριε την υποστήριξή μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ Μαρτίνα. Κάποιοι άλλοι σκιώδεις, συζητητές ή μέλη που θέλουν το λόγο. Και λοιπόν, κάποια κάτι ε, Ευχαριστώ. Αναφέρατε την έρευνα, βεβαίως. Το σύστημα είναι ενιαίο. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμόσουμε τα αποτέλεσματα της έρευνας. Έχουμε μερικές μέρες μπροστά μας για την υποβολή τροπολογιών και βεβαίως θα είμαι σε επαφή με όλους τους κοιόδης συγητές. Πιστεύω ότι οι συνεισφορές από την Επιτροπή μας, από όλους τους ε, σκιωδησίτες, θα είναι απολύτως ε, χρήσιμες για την τελική διατύπωση της γνωμοδότησης. Πρόεδρος, πολύ ενδιαφέρον τομέα για την Επιτροπή μας. Συνάδελφοι, στις 8 ξεκινούμε τις ψηφοφορίες. Βλέπω ότι αποσιάζουν πολλά μέλη τα καλά μέλη, αυτά που συμπαθούν εδώ, ευτυχώ. Θα συνεχίσουμε όσοι είμαστε. Λοιπόν, θα διακόψουμε στο σημείο αυτό ως τις 8 για να ξεκινήσουμε και πάλι με τις ψηφοφορίες. Κύριε Γκρισμπέκ, ξέρω, ξέρω, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε πριν από τις 8. Ε, διακόπτουμε λοιπόν για 10 λεπτά. Ελπίζω να έχω την ανοχή σας. can confirm that we cannot go ahead. Επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε πριν από τις 8. Ο καφές δεν είναι και πολύ μακριά. Λείπαμε για τη διακοπή. Παρουσία του δεν είναι πολύ μακριά. Δεν αστείευομαι. Είναι στα αριστερά σας τα αριστερά μου τουλάχιστον είναι εξαιρετικές. Λοιπόν, ξεκινούμε 8 η ώρα για τις ψηφοφορίες.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 Takie element, no. Element, element. Co? No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 Συνάδελφοι, καθίστε. Καθίστε να αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Καταρχήν να ελέγξουμε ότι όλοι έχουν την κάρτα. Δεν έχετε κάρτα ηλεκτρονική για να ψηφίζετε. Πείτε το μας για να ξέρουμε. Δεν βλέπω να σηκώνει κανεί το χέρι του δεν έχει κάρτα. Υποθέτω ότι όλοι έχουν κάρτα και όλοι είναι εντάξει. Λοιπόν, καθίστε όλοι να αρχίσουμε κανονικά. Θα προσπαθήσω να πάω γρήγορα, ξέρω ότι είναι αργά. Λοιπόν, να τελειώνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πάμε στο σημείο 4 λοιπόν. Ε, σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για εξαίρεση από υποχρέωση θεώρησης για μικρές ε, παραμονές. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ο εισηγητής η εισηγήτρια δεν ζητάει το λόγο. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 45 υπέρ, 2 κατά μία αποχή, συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στην δεύτερη ψηφοφορία. Ε, καταπολέμηση της διαφθοράς και συνέχιση του ψηφίσματος κρίμα. Η Λάουρα Φεράρα είναι η συγγήτρια. Υπάρχει μια, ένα τεχνικό λάθος στο κατάλογο ψηφοφοριών και αφορά το ψήφισμα που αφορά τις τροπολογίες 37 και 38 που δεν καλύπτονται από την τροπολογία 35 και τη συμβιβαστική 2 και θα τεθούν σε ψηφοφορία. Αν αυτό είναι κατανοητό μπορούμε να προχωρήσουμε. Και πριν προχωρήσουμε Θέλω να ρωτήσω τη Λάουρα Φεράρη αν θέλει να μας πει κάτι. Δεν θέλει η Λάουρα Φεράρα. Προχωρούμε κατευθείαν στην ψηφοφορία λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία τροπολογία 14. Ψηφίζουμε. Ένας παραπάνω σοσιαλδημοκράτης ψήφισε. Κύριε Σέκο, δείτε το. Πέρας. Εντάξει και οι σοσιαλδημοκράτες. Δεκτή. Τροπολογία 15. Ψηφίζουμε. Πέρας. δεκτή. 16 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 20. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 22. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 23. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 24. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 26. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Ε, συμβιβαστική 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 34. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 40. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 41. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 43. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 46. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 48. Πέρας. Απερίφθη. 49. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 50 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 3 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 58 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 59 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απερίφθη. 63 ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 64 ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 4 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 5 πρώτο μέρος. θα ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 5, δεύτερο μέρος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. 37. Άρχεται η ψηφοφορία. 37. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 37 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Εψήφισαν όλοι πέρας. Δεκτή 38 ψηφίζουμε. Είπα στην αρχή ότι την 38 θα την ψηφίσουμε. Θυμάστε, μία συνάδελφος θυμάται, άλλος κανείς δεν θυμάται από ό,τι φαίνεται κρίμα. Λοιπόν, 38, ψηφίζουμε ακόμα. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 86 ψηφίζουμε. πέρας δεκτή 110 ψηφίζουμε πέρας δεκτή 111 ψηφίζουμε Πέρας. Δεκτή. Πάω λίγο γρήγορα γιατί είναι πολύ μακρά η ψηφοφορία. Αν θέλετε να επι... τα βραδίνω θα επιβραδίνω. Α, η κυρία ε, ε δεν θέλει να επιβραδίνω. Ψηφίζουμε την συμβαστική έξι άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 108 πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Η 108 τώρα δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 107. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. Η συμβαστική 7 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 57. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 101 ψηφίζουμε. 121 συγγνώμη ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 124 ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 8 πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Ε, συμβαστική 8 δεύτερο μέρος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. 132-133 ταυτόσημες άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτές. 134 ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 135 ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 9 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 138 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 139 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 140. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 141. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 10 πρώτο μέρος ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Συμβαστική 10, δεύτερο μέρος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. 145 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 11 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 151. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 152. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Η συμβιβαστική... Όχι. 161. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 163. Ψηφίζουμε. Πέρας δεκτή 166 ψηφίζουμε πέρας απερίφθη 167 ψηφίζουμε πέρας απερίφθη 168 ψηφίζουμε πέρας δεκτή 169 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 13 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 173 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 179 ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 180 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απερίφθη. 181. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 15 πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 15 δεύτερο μέρος ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 16 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 17 ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 188 ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 189 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 190 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή 191 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή 193 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή 194 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 196. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 197. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 198. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 199 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Η 200 ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. Πάμε στις αναφορικές προτάσεις, τροπολογία 1, ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή η τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 5. Ψηφίζουμε. 5. 5. Τροπολογία 5. Να πάρουμε από το 6 μέχρι το 13 με την αδειά σας όλες μαζί. 5 με 13. Δηλαδή, λοιπόν, 5 με 13 όλες μαζί, αν συμφωνούν όλοι. Όχι. Δεν συμφωνείτε. Εντάξει. λοιπόν, την 5. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 5 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 7. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. Οχτώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτό. 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. Γιατί ποιος δεν ήθελε όλες μαζί. Δέκα. Ε, για να δούμε δέκα. Ψηφίζουμε τη δέκα. Περάς. Δεκτή και αυτή. Έντεκα. Άρχεται την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την έντεκα. Πέρας. Δεκτή. 12 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Και 13 ψηφίζουμε. Κίνγκα πρέπει να ψηφίσεις. Πρέπει. Υποχρεωτικά. Πέρας. Δεκτή και αυτή. 47 υπέρ είναι... κουράζονται και απέχουν λοιπόν πάμε γρήγορα γρήγορα είναι πολλές οι γνωμοδοτήσεις και πρέπει να τις δούμε όλες να πάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα δεν μπορούμε όλες μαζί δεν μπορούμε έχουμε και την ελέγχου προπολογισμών λοιπόν εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Παράγραφος, 2 ψηφίζουμε, Επιτροπή ΔΕΒΕ. Παράγραφος 2. ΔΕΒΕ. Πέρας. Απορριπτεται. Παράγραφος 4 της ΔΕΒΕ ψηφίζουμε. πέρας εγκρίνεται 5 της ΔΕΒΕ ψηφίζουμε πέρας δεκτή παράγραφος 6 της ΔΕΒΕ ψηφίζουμε πέρας δεκτή 8 της ΔΕΒΕ Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. εννέα της ΔΕΒΕ ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. δέκα ΔΕΒΕ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 13 τεβε ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 14 τεβε ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Παράγραφος 5 κοντ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 7 κοντ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 8 Επιτροπή Θεωματικών Υποθέσεων Κοντ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 12 κοντ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 13 παράγραφος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 14 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 18 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 19 ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 19. 20. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 22 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 24 ψηφίζουμε. Πέρασα. Απορρίπτεται. 28. Ψηφίζουμε. 28. 28. Κοντ. Πέρας. Απορρίπτεται. 29. Κοντ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις για την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού υπαριθμών Β αιτιολογική σκέψη ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Αιτιολογική σκέψη Δ, D, άρχεται η ψηφοφορία, recital D. Πέρας. Δεκτό. Δεκτή. Τελική ψηφοφορία Ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 48 υπέρ 3 κατά. Συγχαρητήρια. Στην κυρία Λόρα Φεράρα, την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε πολύ τη Λόρα. Συνάδελφοι, Ερχόμαστε τώρα στη τελευταία ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας, γιατί είναι, παίρνουν χρόνο οι ψηφοφορίες, χρειάζονται πολύ χρόνο. colleagues. Um, Ξεκινούμε λοιπόν με την επόμενη ψηφοφορία που θα κρατήσει και αυτή αρκετά. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και την πειθαρχία σας. Δεν υπήρξαν διακοπές και αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό. Ερχόμαστε λοιπόν στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Παρακαλώ ησυχία συνάδελφοι. Σχέδιο Εκθεση με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η συγκήτρια κυρία Σοφία Ιντβελτ θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε, θέλω να πάρω το λόγο για να ευχαριστήσω θερμά τους όδες εισηγητές, όλους όσοι πρότειναν ε, τροπολογίες του συνεισηγητές ε, στην ΑΦΚΟ αλλά και το προσωπικό το διοικητικό ήταν μια πολύ θετική και επικοδομητική διαδικασία. Η διαδικασία με ικανοποιεί ιδιαίτερως και κατά πάσα πιθανότητα θα με ικανοποιήσει και η έκβαση της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εμείς ευχαριστούμε την Σόφη Ιντφελτ. Με αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ίσως μας πάρει μία ώρα. Ελπίζω να πάμε γρήγορα, όσο δυνατόν πιο γρήγορα και γι' αυτό θα ήθελα την προσοχή σας. Αν είμαστε όλοι ήσυχοι, θα προχωρήσουμε γρήγορα. Αποσύρθηκε η τροπολογία 651. Μόλις μας το είπε η κυρία Χολμάγερ, παρακαλώ σημειώστε το. Ξεκινάμε με τη συμβαστική 16. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 268 ε, ψηφίζουμε τροπολογία 268 Πέρας. απορρίπτεται 270 ψηφίζουμε Πέρας. απορρίπτεται συμβιβαστική 17 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Δεκτή. 283 τροπολογία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή, δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 284 άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, λέει η γραμματεία. Δεν το ψηφίζουμε. Ζήτω συγγνώμη συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη και πάλι. Έχουμε προφορική τροπολογία από την κυρία Σπινέλη πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο υπάρχει αντίθεση στην προφορική τροπολογία της κυρίας Πινέλη. Εάν δεν υπάρχει, τι ψηφίζουμε. 2.84 ψηφίζουμε τώρα. Ζήτω συγγνώμη, δεν ήμουν ενημερωμένο. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 2.88 ψηφίζουμε. Όχι, 285 καταπίπτει. Είμαστε στη 288 και ψηφίζουμε. Τώρα ξεκίνησε το μηχάνημα. Ψηφίζουμε τη 288. Στο συγγνώμη για την καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος. Πέρας. Απορρίπτεται. 289 ψηφίζουμε. Να κάνουμε τη 289 πάλι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.90 προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε. Πέρασε. και τα μηχανήματα κουράζονται. Συμβιβαστική 18 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. Τροπολογία 2.95. Ψηφίζουμε. Πέρας. δεκτή. 2.96 ψηφίζουμε. Πέρασα. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασα. Δεκτή. Συμβιβαστική 19α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 3.11 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογική. Συμβιβαστική 20. Όχι, εγκρίθηκε, το συγγνώμη. Τροπολογία 321. Τροπολογία 321 ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 322 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.23 και 3.24. Ψηφίζουμε μαζί την είναι ταυτόσιμες. Πέρας. Απορρίπτονται. 3.27. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 328. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 329 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.40 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.41-3.42 ψηφίζουμε μαζί, είναι ταυτόσιμες. Πέρας. Απορρίπτονται. 3.46 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία 22, πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 370. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 3.99. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 400 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 402. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. ψηφοφορία ε, σε ομαδική. Τροπολογίες 23 31, 36, 43, 45, 48, 52, 54, 58 και 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε μαζί. Πέρας. Δεκτές. Τροπολογίες 5 και 4. 4. Ψηφίζουμε την 4. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 7. Πέρας. Απορρίπτεται. 8. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 9. Ψηφίζουμε. Πέρας. 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 11, τροπολογία 11. Την τροπολογία 11. Ναι, συναδελφοί, την τροπολογία 11 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 15. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Πέρας. Απορρίπτεται. 18. Πέρας. Απορρίπτεται. 19. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 20. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 21. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 32-35 είναι ταυτόσημες. άρχεται η ψηφοφορία για την αιτιολογική αναφορά 11. Πέρας. Απορρίπτεται. 37 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 38 ψηφίζουμε. Close. Πέρας. Απορρίπτεται. 39-40 ταυτόσιμες έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 42 έναρξη ψηφορίας πέρας απορρίπτεται 46 άρχεται πέρας απορρίπτεται 47 άρχεται πέρας απορρίπτεται 53 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 59 άρχεται. Πέρας. Ψηφορίες. Απορρίπτεται. 661, 61, 62, 63. Ταυτόσιμες άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Αποδεκτή. 66 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 67 και 68 ταυτόσημες άρχεται η ψηφορία. Πέρας εγκρίνεται 69 άρχεται όχι λέει ο πρόεδρος όχι 69 70 για αποσυρθεί 69 71 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 72 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 73 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 74 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 75 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 83 ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορία συγκρίνεται 88 ψηφίζουμε. Πέρας απολύτεται 89 ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται 90 και 91 ταυτόσημες ψηφίζουμε. Πέρας. ψηφοφορία Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Ψηφίζουμε. Πέρα. Εγκρίνεται. 96 ψηφίζουμε. Πέρα. Είστε, είστε καλά, ελπίζω εγκρίνεται. Αφού ψηφίσετε όλα καλά, 97 ψηφίζουμε. 97, θα παραλαμβάνω Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 105. 105 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 106 ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφορία συγκρίνεται. 118. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφορίας. Εγκρίνεται. 133 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται συμβαστική 7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 139 ψηφίζουμε. πέρας απορρίπτεται 141 ψηφίζουμε πέρας ψηφορίας εγκρίνεται συμβιβαστική 9 ψηφίσμα. πέρας εγκρίνεται 147 άρχεται η ψηφορία. Πέρας ψηφορία, απορρίπτεται 148 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 149 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 161 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 173 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 174 ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 175 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας εγκρίνεται 176 ψηφίζουμε πέρας ψηφορίας απορρίπτεται 177-178 μες ψηφίζουμε πέρας ψηφορίας απορρίπτεται 179 ψηφίζουμε Πέρας. Ψηφορίας. Απορρίπτεται. 180. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 183. Ψηφίζουμε. Πέρας απορρίπτεται. 184 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 185 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 186 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 187. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφορίας. Εγκρίνεται 188. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Ψηφορίας. Απορρίπτεται 189. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική 12 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας εγκρίνεται 199 και 200 ταυτόσιμες ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται, απορρίπτονται. 201, ε, 2 και 3 ταυτόσιμε ψηφίζουμε. Πέρας ε, ψηφορία απορρίπτεται. 204, 205 και 206 ταυτόσιμες ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτονται. 209 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορές απορρίπτεται. 2.07 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 210 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας απορρίπτεται. 211 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας απορρίπτεται. 208 άρχεται η ψηφορία. Πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 221. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 2-2-2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφοφορίας εγκρίνεται 223. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Ψηφοφορίας εγκρίνεται 224. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται. 2.25 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. 2.45 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. 2.50 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.52 Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 253-254 ταυτόσμες. Όχι, λέει ο πρόεδρος. 253-254 ψηφίζουμε. Πέρας απορρίπτεται. 2.55 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.56 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Όχι, με email δεν δεχόμαστε ψήφους. Απορρίπτεται. Λοιπόν, ε, και εδώ μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα, έτσι. Δεν γίνεται με email. Οπότε πάμε στο παράρτημα, λεπτομερείς συστάσεις. 404. ψηφιζουμε Πέρας Πέρασε ψηφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3α. Ψηφίζουμε. πέρας απο από ψηφοφορία. 3 συμβαστική ψηφοφορια ψηφοφορίας έναρξη συμβιβαστικη Πέρασε. Εγκρίνεται συμβαστική. Αμεσούρετε 4-6-3. 4-6-3 Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Ψηφίζουμε. Με συγχωρείτε. Συνάδελφοι. Ε, πριν από αυτό έχουμε την 464. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 464. Ψηφίζουμε ακόμη. Πέρασε. Ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. συμβαστικη 4. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 6. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Καλά νέα. Ε. ε συμβαστική 8. Πιάνει μια ολόκληρη σελίδα. Μέσα στην τελική ευθεία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβαστική 10 ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβιβαστική 11 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 629 και 630 ταυτόσημες ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Έξι τριάντα ένα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.42 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας, Απορρίπτεται. 6.41 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 6.40 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 6, ναι, με 13 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. 647 ε, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Rejected. Απορρίπτεται 648 ψηφίζουμε. Πέρας. 649 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 6.50. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεκτή. 6.52. 51 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε την 6.52. Πέρασε. Δεκτή. 6.53 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 654 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Αναφορικές προτάσεις σε αιτιολογικές σκέψεις. Άρχεται η ψηφοφορία 305. Όχι. Όχι, στη, όλες μαζί. Όλες μαζί θα είμαστε εκεί που είναι όλες μαζί. ε, όλες μαζί τις ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, δεν... Ε, ε, ε ήθελα να δω ε, τι προσέγγιση έχουμε ε, ως ομάδα. Λοιπόν, 408 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 409. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 411. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 413. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 4-14 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 4-15 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 4-20 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 421. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 422 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 423 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 4, 25, 26 μαζί ψηφίζουμε. Είναι ταυτόσιμες. Πέρας. Δεκτές. 4, 27, 24, 28 ψηφίζουμε. Είναι ταυτόσιμες και αυτές μαζί. Πέρας. Δεκτές. 4, 29 Α, όχι. Ήτανε, ήτανε και αυτή έπρεπε να πάει. Ε, 3-3-1, 3-3-3-2. Ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Δεκτή. 4-33 ήταν τελευταία. Ε, ναι. Και 4-34-4-35 ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Τι, να ξαναψηφίσουμε οι 434 και 435 ταυτόσιμες ε, είχαμε τελ... ξαναψηφίζουμε. Είχαν να γίνει δεκτές. 436, 437 ταυτόσιμες ψηφίζονται. Πέρας. Απορρίφθηκαν. 440 ψηφίζουμε. Πέρας. Εμείς τώρα είμαστε στις 4.40. Άρχεται η ψηφοφορία 4.40. Μα το ή, μα την ψηφίσαμε, δεν την ψηφίσαμε. Τι κάναμε. Πέρας τέλο πάντων στην 4.40. Απορρίπτεται. Φαίνεται 441. Ψηφίζουμε. 441 ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. 442 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 443 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 444 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 445 ψηφίζουμε. Τελειώνουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 446 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 4.47 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 4.48 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 4.49 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 454 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στη γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ. ΑΦΚΟ 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. ΑΦΚΟ 9. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. ΑΦΚΟ 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Αύκο 13 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Αύκο 14 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται αυτή. Αύκο 18 ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. Και πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία που θα γίνει ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία, συνάδελφοι. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή 49 υπέρ, 11 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας, ήταν μακρά η ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες, τελειώσαμε και τη συνεδρίαση, αν δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ανακοινώσω μία ψήφο μειοψηφίας. Υπάρχει με βάση τον κανονισμό 56 της γραπτής διαδικασίας, ε, είναι γνωστό εντάξει.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 θα υποβάλουμε και θα δημοσιεύσουμε ε, έκθεση αντίθετη προς αυτή διότι έτσι πιστεύουμε ότι θα παρακάμπτονται ευρωπαϊκές συμβάσεις και συνθήκες. Ε, μπαίνουμε δηλαδή σε χωράφια που είναι του Συμβουλίου με βάση το κανονισμό, το άρθρο του κανονισμού 56, μπορεί να ε, ε, υπάρξει ε, μέχρι 200 λέξεις μία δήλωση της μειοψηφίας. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό, προβλεπόμενο και οι δύο συνάδελφοι είπαν ότι θα το κάνουν. Αυτό μπορεί να γίνει και μπορεί να ψηφιστεί μια τέτοια γνωμοδότηση αν τεθεί σε ψηφοφορία και θέλουν. Αν δεν υπάρχει τίποτε στα διάφορα, κλείνω τη συνεδρίαση. Ναι, μπορείτε, έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό, να κάνετε δήλωση μειοψηφία ε, με βάση το άρθρο 56 του κανονισμού και τώρα αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο, κλείνουμε τη συνεδρίαση.